Συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας ε, της ε, Επιτροπής Βιομηχανίας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους ε, θερμά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα καινούργια πρόσωπα που βλέπω και τους εύχομαι σε όλους να έχουμε μια καλή συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας ε, επισημάνω ότι η Επιτροπή μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα με τις κάμερες. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι σας ε, γνωρίζετε το στόχο της ε, συνεδρίασής μας. Ε, σήμερα πρέπει να συστήσουμε το Προεδρείο της Επιτροπής μας με την εκλογή του Προέδρου και τριών αντιπροέδρων σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού. Θα εκλέξουμε ή 181 με συγχωρείτε. Πρώτα θα εκλέξουμε ε, τον πρόεδρο και μετά τους αντιπροέδρους. Ε, προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας ε, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την εκλογή του πρόεδρου. Σύμφωνα με τον 95 κάθε, παράγραφος 2 χρειαζόμαστε για να έχουμε απαρτία το 1 τέταρτο των μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας. θεωρώ λοιπόν ότι ασυζητητή διαθέτουμε απαρτία. Και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να καταθέσετε τις προτάσεις για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Βιομηχανή. Η κυρία Ντεκαστήγιο έχει το λόγο. Τον κύριο Ρολ θα ήθελα να προτείνω για πρόεδρο. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Herbert Ρόιλ ε, προτείνεται για τη θέση αυτή. Αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση, διαβοής ε, εκλέγουμε τον ε, νέο πρόεδρο. Ε, συνάδελφε κύριε Ρόιλ, ε, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ θερμά για την εκλογή σας, να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ στο βήμα και ε, το διαδικαστικό του κυρίου Τόρμες φαντάζομαι θα το ρυθμίσετε εσείς, έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία λοιπόν, ελάτε εδώ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν όμως πω και εγώ κάτι, ο συνάδελφος κύριος Τούρμες ζήτησε το λόγο επί διαδικαστικού και σε εκ τούτου προηγείται. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την ανάληψη αυτής της τόσο σημαντικής θέσης. Και εδώ ως πράσινη, εδώ και χρόνο εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούμε να σας πείσουμε να μας πείτε κατά πόσον μέσα από αυτή τη θέση που αναλάβετε θα προωθήσετε τις δικές σας τις θέσεις, τα δικά σας συμφέροντα ή αυτά που έχουμε συμφωνήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Ας πούμε για τα κτίρια, για την ετικετοθεσία. Για μας όλους είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε μερικά λόγια επ' αυτού, να μας πείτε πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε αυτή τη θέση του Προέδρου τη στιγμή που ε, θα συμμετέχετε συμμετέχετε στο μέλλον σε τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, τόσο σημαντική σας ερώτηση. Άλλο διαδικαστικό παρακαλώ. Κοιτάξτε, σύντομη παρατήρηση και εγώ βεβαίως ε, πρώτα απ' όλα σας συγχαίρω θερμά και προτείνω ο νεοεκλεγής ε, πρόεδρος να είναι εξίσου αντικειμενικός όπως ο συνάδελφος κύριος ε, Τόρμες για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί σας είχαμε κύριε Τούρμες ως εισηγητή και ξέρουμε πολύ καλά να κρίνουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά λοιπόν από αυτά τα πολύ χαρούμενα και ευχάριστα <laughs> σχόλια, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ, αλλά με συγχωρείτε πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκούμπελς. Αγαπητέ Πρόεδρε, και εγώ ε, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και να σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ε, για τη δουλειά που θα κάνετε. Και να ε, ξεκαθαρίσω, εγώ δεν συμμερίζομαι και δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Τούρμες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Εξ ονόματος της ομάδας μας, ε, των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Γνωρίζω τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε. Καλή τύχη. Ο κύριος ε, Χατζημαρκάκης, ε, ε, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Ρόλ, και εμείς οι φιλελεύθεροι δημοκράτες αυτού του σώματος θα θέλαμε να σας συγχαρούμε, να σας ευχηθούμε βόδες των εργασιών σας και γνωρίζετε πολύ καλά, το παν στη, στο Κοινοβούλιο είναι η διαφάνεια. Να, παρακαλώ εσείς. Ο κύριος Χαντστόφ. Αξιότιμε κύριε Ρόιλ, εγώ στηρίζω την εκλογή σας και πρέπει να πω ότι στην Επιτροπή μας ε, συμπεριφερθήκατε πάντα με μεγάλη αξιοπρέπεια. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι είμαι κατά ε, των, ε, της δυσφήμισης ε, που έχετε υποστεί στο πρόσωπό σας. Η κυρία Ουλάφσκακοκ ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Ουλβ Κούκε είναι η σωστή προφορά. Ε, θέλω να πω και εγώ ότι ως ε, Αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ είμαι νεοεκλεγήσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαια προφανώς και νέο μέλος της Επιτροπής ε, Ήτρα και ελπίζω ότι θα έχουμε επικοδομητικές, έστω και σκληρές ενίοτε συζητήσεις. Εμείς λοιπόν στην ομάδα μας προσβλέπουμε σε πολλές ε, συζητήσεις, αποφάσεις ε, μεγάλης ε, σημασίας σε αυτήν την Επιτροπή κατά τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σα. Παρακαλώ. Εξ ονόματος ε, της ε, Γκουέ θα ήθελα να σας συγχαρώ. Ονομάζομαι Ματίας. Ε, σας εύχομαι καλή δουλειά. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε όλοι μαζί. Επικοδομητικά. Καλή δουλειά σε όλους. Thanks. So, meine lieben Kollegen... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω για άλλη μια φορά. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ θερμά που με εκλέξατε σε αυτή τη θέση. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αποτελεί διάκριση για μένα και βεβαίως και ένα σοβαρό καθήκον. Πολύ μεγάλη η ευθύνη, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε μια επιτροπή που έχει μεγάλη σημασία, που είναι δύσκολη, είναι μια επιτροπή ε, που έχει να αντιμετωπίσει πολλές ε, πολιτικές αντιπαραθέσεις, κάτι το οποίο είναι καλό και σωστό για τη δημοκρατία. Εξάλλου είναι και μια επιτροπή που έχει μια πολύ καλή παράδοση με την κυρία Αγγίλικα Νίπλερ. Ε, προφανώς είναι δύσκολο να είναι κανείς διάδοχός της. Πάντως σας ευχαριστώ θερμά και για ένα πράγμα μπορείτε να είστε σίγουροι. Εγώ θα εργαστώ με τέτοιο επαγγελματισμό που είναι ο απολύτως απαραίτητος. Δίκαια, όπως ακριβώς καλείται να το πράξει ο πρόεδρος μια τέτοια επιτροπή. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν έχει καμία σημασία το ότι προφανώ όλοι μα έχουμε ίσω ε, τι δικέ μα προσωπικέ απόψει και διαφορετικέ. Μα αυτό είναι και το ωραίο στη δημοκρατία, το ότι μπορούμε να εκφραστούμε. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και το κέρδο τη Νέα Ευρώπη. Ότι μπορούμε σε όλα τα κράτη τη Ευρώπη να δεχόμεθα διαφορετικέ απόψει, να δεχόμεθα την πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ ω πρόεδρο, φέρω ε, τεράστια ευθύνη το γνωρίζω ε, και πρέπει να ξέρετε ότι θα ανταποκριθώ σε αυτήν. Ως Επιτροπή ε, φέρουμε και άλλη μια μεγάλη ευθύνη μετά από αυτές τις ευρωεκλογέ, όπου είδαμε ότι οι πολίτες δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένοι. Το κατά πόσον είμαστε αποτελεσματικοί, κατά πόσον παρουσιάζουμε προγράμματα τα οποία πείθουν τους ανθρώπους ότι έχει νόημα να υπάρχει η Ευρώπη, αυτό θα αποδειχθεί μέσα από την καθημερινή μας εργασία, αποτελεί πρόκληση για όλους μας και ελπίζω να ανταπεξέλθουμε όλοι από κοινού να αντιμετωπίσουμε σημαντικά θέματα που ε, θα έχουν πολλές αντιπαραθέσεις. Ελπίζω λοιπόν στα σημαντικά αυτά θέματα να βρούμε και το χρόνο να προχωράμε σε βάθος που σημαίνει ότι σε επουσιώδη ζητήματα θα πρέπει να προχωράμε λίγο πιο γρήγορα έτσι ώστε στα πραγματικά ουσιώδη να έχουμε το χρόνο και να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες και επιπλέον ως Επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου και σε άλλε προκλήσει, Συμβούλιο, Κομισιόν, άλλε επιτροπέ που έχουν διαφορετική άποψη, να μπορούμε να σταθούμε. Εμεί ε, δεν είμαστε θηγατρικοί καμία επιτροπή. έχουμε δικά μα ε, θέματα, βιομηχανία, έρευνα, τεχνολογία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα συμφέροντα γενικότερα που υπάρχουν στην κοινωνία. Σε οικονομικά χαλεπούς ε, καιρού. Εμεί καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε μια ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη και είμαι σίγουρος ότι θα ανταπεξέλθουμε στο καθήκον μας. Εγώ ό,τι μπορώ να κάνω θα το πράξω. Σας παρακαλώ όλους να με συνδράμετε και τους παλαιούς και τους νέους και όλα τα πολιτικά κόμματα. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι αγαστή συνεργασία ανάμεσά μας και με τα μέλη της γραμματείας που τα χρειαζόμαστε για να παρουσιάσουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ και όπως σας είπα εύχομαι καλή συνεργασία. και πάμε τώρα, αν θέλετε, στο επόμενο θέμα όπου ε, εκλέγουμε τους αντιπροέδρους. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων να καλύψουμε. Τα ονόματα, μισό λεπτό, Προτείνουμε λοιπόν το Ρούντε, ποδηματά και, μισό λεπτό, και του Ζινόφσκι. Επιθυμεί κάποιος άλλος ε, να καταθέσει άλλη πρόταση για τις, τους αντιπρόεδρους. Από ό,τι βλέπω όχι. Τώρα πώς θα γίνει, θα πρέπει να ψηφίσουμε για κάθε ένα ξεχωριστά ή μήπως μπορούμε να το διεκπαιρώσουμε συλλήβδιν. Το θέμα έληξε, συμφωνήσατε διαβοής και οι τέσσερις αντιπρόεδροι εκλέγονται. Ε, τους συγχαίρω και τους παρακαλώ να έρθουν εδώ να κάτσουν στο βήμα έτσι ώστε για τρία-τέσσερα λεπτά να διεκπαιρώσουμε κάποια διαδικαστικά κυρίως το κατά πόσον την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουμε ή όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ε, τα επίσημα τα διεκπαιρεώσαμε, τώρα πλέον μπορούμε να αναλάβουμε το έργο μας. Ε, έχουμε λίγα λεπτά. Η γραμματεία μου επισήμανε ότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσον την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουμε ή όχι. Αν θέλουμε μπορούμε και να μην συνεδριάσουμε. Η Επιτροπή λοιπόν με βάση ε, το πρόγραμμα των συνεδριάσεων ε, μπορεί να συνεδριάσει από τις 9 μέχρι τις 12.30 το πρωί. Τα θέματα για την Επιτροπή μας είναι τα εξής. Πρώτον, να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τα επίγοντα και για τα θέματα που εκκρεμούν. Θέλω όμως να πω, ένας άλλος βασικός λόγος γιατί πρέπει να συνεδριάσουμε και νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, ε, πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι συντονιστές, είναι το θέμα της οργάνωσης των εργασιών μας. Παραδείγματος χάρη, τον Οκτώβρη, πότε θα συνεδριάσουμε, γιατί η κατάσταση με την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής ε, δημιουργεί κάποιες ε, αναβολές μεταθέσεις το χρόνο. Άρα πρέπει να είμαστε λιγάκι συγκεκριμένοι. Δεύτερο ερώτημα που πρέπει να διευκρινιστεί. Κατά πόσον θα πρέπει να ε, δεχθούμε ή να υποβάλουμε προσκλήσεις στη Σουηδική Προεδρία και τρίτο θέμα τι θα κάνουμε με τους ε, τρεις ε, φακέλους ε, που τρέχουν, που είναι εν Είναι οι φάκελοι εκείνοι που βρίσκονται στην έχουν περάσει την πρώτη ανάγνωση και πρέπει να αποφασίσουμε αν θα περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση και επειδή είναι πολλοί νέοι συνάδελφοι κατά πόσο πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτά είναι τα θέματά μας και γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε. Θα, θα συνεδριάσουμε την επόμενη εβδομάδα φτάνει η Επιτροπή των Συντονιστών ή τα θέλετε και τα δύο. Παρακαλώ να πείτε τώρα τη γνώμη σας για να σχηματίσουμε άποψη, γιατί δεν θέλω να αποφασίσω μόνος μου. Λοιπόν, πρώτος που ζήτησε το λόγο είναι ο συνάδελφος κ. Τσίτσεστερ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν Είμαι υπέρ του να έχουμε συνεδρίαση της ε, Επιτροπής, που ίσως είναι κάπως νωρίς, αλλά χρειάζεται σίγουρα συνεδρίαση των συντονιστών. Και θα ήθελα να προτείνω και μάλιστα να κάνω ένα αίτημα να γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών πρώτα, το πρωί της Τρίτης, ώστε οι συντονιστές να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα διάφορα που θίξατε και οποιοδήποτε άλλο θέμα θα έχει προκύψει μέχρι τότε. Μάλιστα να σας πω ότι πολλοί συνάδελφοι είναι έτοιμοι να πάνε πια διακοπές. Και δεν θέλω να τους εμποδίσουμε ε, κάνοντας μια ε, συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα μπορούσε να περιμένει για μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Συμφωνώ με τον κύριο Τσίτσεστερ 100%. Πώς θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Περάσαμε μια ολόκληρη θητεία δίπλα-δίπλα, εργαζόμενοι μαζί. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη θεωρεί πως ε, δεν χρειάζεται να ε, συγκαλέσουμε την Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ίσως όμως ε, χρειάζεται οι συντονιστές να, να βρεθούμε μεταξύ μας μια πρώτη φορά, γιατί πράγματι πριν φύγουμε για διακοπές θα πρέπει να προετοιμάσουμε την ε, πρώτη συνάντηση της Επιτροπής ε, το Σεπτέμβριο. Συμφωνώ λοιπόν πλήρως με τον κύριο Τσίτσεστερ. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Θα συνεργαστούμε σίγουρα πολύ καλά και συμφωνούμε κι εμείς ως ομάδα ότι θα ήταν υπερβολικά βεβαιασμένο να κάνουμε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στην ε, Βρυξέλλες, καλύτερα μια συνάντηση των συντονιστών. Ε, äh, Ο κύριος Χατζημαρκάκης, ε, πρόεδρε, συμφωνώ με τον κύριο Τσίτσεστερ που είπε ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε συνεδρίαση συντονιστών. Πρέπει όμως ε, να πούμε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τη διαδικασία της ε, πρώτης ανάγνωσης. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι συνάδελφοι. Ε, μπορούμε λοιπόν την ίδια ημέρα να έχουμε έτσι μια σύντομη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να έχουμε μια σύντομη διάρκεια συνεδρίας Επιτροπής. Ο κύριος Τούρμες, κατά κανόνα, συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Χατζημαρκάκη, αλλά Τώρα η άποψη του κυρίου Τσίτσεστερ είναι πιο σωστή. Ε, την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μόνο συνεδρία συντονιστών, όχι επιτροπή, είναι πολύ νωρί ακόμα. Και εξάλλου, ε, και επειδή πολλοί από εμά κουραστήκαμε στι ευρωεκλογέ, ε, να έχουμε άλλη μια εβδομάδα ε, διακοπέ. Το όνομά σα, παρακαλώ, δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σα. Ο κύριο Βασκό. Σα ζητώ συγγνώμη, με τα ονόματα λιγάκι δεν τα πάω ακόμα καλά. Θα τα μάθω όμω. Ε, θα τα μάθω και δεν βλέπω και μακριά. Ο συνάδελφος Βάσκο. Μπόλτσο λέγομαι και είμαι από την Ουγγαρία. Είμαι στους μη εγγεγραμμένους. Ε, πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε αντιπροσώπευση σε αυτή την Επιτροπή μέχρι τώρα και τώρα θα είμαι ο συντονιστής των δύο μη εγγεγραμμένων μελών. Αλλά θα ήθελα ε, να λάβω και όλη την τεκμηρίωση την οποία αναφέρατε, τα έγγραφα της πρώτης, ανά, της πρώτης ανάγνωσης κτλ. Έτσι ώστε να προετοιμαστώ έστω για τη συνάντηση των συντονιστών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι η Γραμματεία προφανώς θα σας ε, βοηθήσει. Αυτό αφορά όλους τους συναδέλφους που είναι νέοι. Ε, βεβαίως ε, είναι σαφές ότι δεν ξέρετε τι έχει προηγηθεί. Ανακεφαλαιώνω σύντομα. Αν κατάλαβα καλά, στην κύριε Χατζημαρκάκη, εφόσον συμφωνείτε και εσεί. Ε, οι περισσότεροι λένε ότι δεν είναι απολύτω απαραίτητο να έχουμε την επόμενη εβδομάδα συνεδρία τη Επιτροπή. Συμφωνείτε επ' αυτού να μην συνεδριάσουμε την επόμενη εβδομάδα ω Επιτροπή, αλλά να συνεδριάσουν οι συντονιστέ να προετοιμάσουν τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Προτείνω λοιπόν ε, οριστικά πλέον θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα οι συντονιστές και δεν θα συνέλθει η Επιτροπή. Η κυρία Ματίας έχει το λόγο. Να επιβεβαιώσω και ότι από πλευρά μας η ομάδα μας συμφωνεί με το να γίνει μόνο συνεδρίαση των συντονιστών και ότι η συνεδρίαση της, ομάδας, τη Επιτροπής σε πλήρη σύνθεση να γίνει μετά τι διακοπές. Πολύ ωραία λοιπόν. Την επόμενη Τρίτη το πρωί οι συντονιστές, η Επιτροπή μετά τις διακοπές και τα θέματα θα στήσουμε είναι οι ημερομηνίες, οι φάκελοι, τα θέματα δηλαδή και η πρόσκληση από και προς τη Σουδική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεδρίαση. Όσοι δεν έρθουν εδώ την επόμενη εβδομάδα τους εύχομαι καλές διακοπές. Τις κερδίσανε με το σπαθί τους όλοι και όσοι δεν θα φύγουν την επόμενη εβδομάδα θα φύγουν λίγο αργότερα. Γεια σας.